Ευρωπαϊκή Ένωση την Ουκρανία. Νομίζω ότι η ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγικό μα στόχο και θα πρέπει να βρούμε τα δειγμένα μέτρα για να φτάσουμε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ανδρίκενα και ακολουθεί ο κ. Μίλσκι.